Good afternoon, colleagues. Καλό σας απόγευμα, συνάδελφοι. Έχει περάσει η ώρα. Καθίστε. Μην προσδεθείτε, αλλά θα ήθελα να αρχίσουμε παρόλα αυτά. So, welcome to, to this. Uh, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας, στην απογευματινή συνεδρίαση και θα ψηφίσουμε καταρχήν στο σχέδιο γνωμοδότησης για τη βελτίωση πρόσβασης σε φάρμακα και θα ήθελα το ταχύτερο δυνατόν να αρχίσουμε. Okay. Compromise amendment number one. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε. Την 5 ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας και εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. αυτό ήταν το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 19. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 29. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της συμβαστικής 5. Πέρας εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε λοιπόν την 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται να ελέγξουμε την 52, ελέγχουμε την 52. Απορρίπτεται. Συμβασμός 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Την παρέλειψα υπέρ της 56, 56 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 59 τώρα, 59. Ψηφίσαμε τη συμβαστική 7. Τροπολογία 59 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά αποχές ναι καταπίπτει με συγχωρείτε 57 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε την 57 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, πρέπει να ελέγξουμε, πρέπει να ελέγξουμε. Συμβιβαστική τροπολογία 10, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με δύο ψήφους παραπάνω. 92. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ Κατά. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Ε, δεύτερο τμήμα της 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. Εντάξει. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, και πάλι πρέπει να ελέγξουμε. 95 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε και πάλι. 54 αρχίζει ο έλεγχος. Πέρας εγκρίνεται κατά μία ψήφο. Σι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα τελική ψηφοφορία στο σχέδιο ψηφίσματος, στο σύνολό του, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Τώρα προχωράμε στην ε, δεύτερη ψηφοφορία. I have it, and I hope I hear. Sorry. Okay, we continue with the annual report of the activity. Συνεχίζουμε λοιπόν με την έκθεση για την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή κατά το 2015. Σεμιβαστική α, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 14, υπέρ. Δεύτερο τμήμα μόνο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας για την Β1. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η Β2, συμβιβαστική Β2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 24, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 25, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26, υπέρ. 26 και 27, καθώς είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Έλεγχος. Έλεγχος να λέτε. Όχι, όχι. Είναι πιο ευγενικό. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, λοιπόν. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ε, εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Έλεγχο ζητείτε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C1. Υπέρ. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε μπερδευτεί λόγω τη εκλογή του Τραμπ, λέει η πρόεδρο. Υπέρ λοιπόν για τη Σιένα. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Η C2, παρακαλώ. Συμβαστική C2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έγκρινεται. 30. Μισό λεπτό. Η 35. Για στι δύο ζητείτε παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Με τεράστια διαφορά εγκρίνεται. 35 τώρα παρακαλώ. Και 36 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία D1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική D2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζητείτε έλεγχος για τη συμβιβαστική D2. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 43. Πέρας. Εγκρίθηκε. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Γιατί δεν σηκώνετε καλά τα χέρια σας βασικά. 49 παρακαλώ. Έλεγχος. Πέρασε. Πενήντα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται 60 υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται 61 υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία G. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ζητείτε έλεγχος για την G, παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας τώρα. Απορρίφθηκε. Και τώρα πάμε στην τροπολογία υπαριθμών. Α, όχι, έχουμε να ψηφίσουμε τις μεμονωμένες τροπολογίες. 66 παρακαλώ. Και 67 ταυτόσιμες. Όχι, ξεχωριστά τι θέλετε. 66, υπέρ. Είναι ταυτόσιμες. Είναι εντελώ ίδιες. Άρα θα τι ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έστω για την 66 και την 67. Πέρας. Απορρίπτονται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 42. ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρας. Εγκρίθηκε με μία ψήφο. Διαφορά. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ χρειάζεται έλεγχος για την 72. Έναρξη παρακαλώ. Της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη τελική σκέψη, 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Τέσσερα παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. Πέντε υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. Έξι υπέρ. Okay. Okay. Let's be, let's be... Μάλιστα, για να είμαστε πολύ ευγενείς προς το ΕΛΚ. Να είμαστε πολύ ευγενεί στους συντονιστέ. Θέλετε ένα λεπτό, πέντε λεπτά, πόσα θέλετε. Σχόλια το μικροφόνο. Να κάνουμε μια δημιουργική παύση, όπω λένε και στην τηλεόραση. Θέλει κανεί ε, να μα πει κανένα έκδοτο, να μα τραγουδήσει κάτι. Να γεμίσουμε την ώρα μα. Can I, just... Sorry, but it is unusual. Κοιτάξτε, είναι λίγο ασυνήθιστο να διακόπτονται οι ψηφοφορίε. Ξεκινήσαμε, ας συνεχίσουμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Και το ΕΛΚ να ακολουθήσει το συντενιστή του. Να προχωρήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι τα διευκρινίσαν τα όσα είχαν να διευκρινίσουν, λέει η Πρόεδρο. Τώρα να, ψηφίσουμε την 6, τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκριθήκε. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έλεγχος για το πρώτο τμήμα της 9 παρακαλώ. Έναρξη ψηφορίας. And the vote is closed. Πέρας, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 9, ε, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 10, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 11. Με νέα τροπολογία, προφορική. Όπως βλέπετε στο κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκριθήκε. Η 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Έλεγχος για τη 15. Ελέγχουμε τη 15. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Η 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να άλλαξουμε παρακαλώ και τη 16. Έναρξη ψηφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου έκθεσης, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρασε. Εγκρίθηκε. So, thank you every... Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε, που φέρατε και τις ε, κάρτες ψηφοφορίας. Το επόμενο θέμα αφορά τη γνωμοδότηση σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Can I have, uh, can you pass to the next subject, please? Just, which opinion you're talking about? Σας έδωσα το λόγο ως εισηγητή για το επόμενο θέμα, κύριε Μαριά. Έχετε το λόγο. This time I need a break. <laughs> Τώρα το χρειάζομαι το διάλειμμα. Thank you, Madam Chair. Uh, can I use this time for a very short statement on behalf of the EPP Group to the... Πρόεδρε, να κάνω ένα σχόλιο εξ ονόματος του ΕΛΚΑ, μιας και έχουμε λίγη ώρα. Αγαπητή Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας του ΕΛΚΑ θα ήθελα να πω το εξή. Η πρώτη ψηφοφορία για την γνωμοδότηση για τι επιλογέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την βελτίωση τη πρόσβαση σε φαρμακά ήταν σημαντικό έγγραφο, αλλά δυστυχώ. Uh, Στην τελευταία φάση της προετοιμασίας του κειμένου, θεωρώ ότι δεν υπήρξε ιδέουσα σοβαρότητα. Γι' αυτό δεν ήταν ικανοποιημένη η ομάδα του ΕΛΚ Και γι' αυτό τελικά αναγκαστήκαμε, χωρίς να το θέλουμε, να καταψηφίσουμε. Αυτή είναι η θέση του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόεδρος. Έτσι έχει η δημοκρατία. Το σημειώσαμε και περνάμε στην επόμενη, στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη γνωμοδότηση. Δεν ξέρω, ο κύριος Μαριάς ε, τα βρήκε, είναι έτοιμος. Okay, then we, we do this without your contribution. Κοιτάξτε, τώρα θα το κοιτάξουμε το θέμα χωρίς να σας ακούσουμε. Θα σας δώσω και το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα εξετάζεται την τροπολογία αυτή και ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το και καιρό. Προθεσμία καταθέση τροπολογιών 21 Αντεκάτου και θα ψηφίσουμε στις 24 στην Επιτροπή, 24 Πρώτου. και μετά στην Ολομέλεια. Ο κύριος Μαριά δεν είναι σε θέση να πάρει το λόγο. Κανείς από τους κοιόδη θέλει να πάρει το λόγο. Αν όχι. Α, εφόσον ζητάτε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σεσίλια. Είναι λίγο περίεργο να σχολιάζουμε μία γραμματοδότηση, τον δεν έχουμε καν ακούσει τον εισηγητή. Αλλά εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα θέλαμε παρόλα αυτά να πούμε ότι θεωρούμε ότι είναι ένα σαφέ σημείο αυτή η γνωμοδότηση. Αποτελεί μία βάση για να ακουστεί η φωνή των πολιτών για την ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη ρυθμίση. Ένα γενικό σχόλιο από πλευρά μα ότι η καλύτερη ρύθμιση για μα αφορά την βελτίωση του νομοθετικού συστήματο και του συστήματο νομοθεσία δεν είναι εφημισμός για να καταργούνται δικλείδες ασφαλείας για τα δικαιώματα των πολιτών και των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν να αποτελεί μια ευκαιρία για να κοιτάμε το πώς μπορούμε να ε, ληφθούν καλύτερα υπόψη τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στην διαδικασία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προκειμένου να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση στη νομοθεσία. Και έτσι λοιπόν εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε ότι η διαδικασία νομοθεσία και του νομοθετικού έργου δεν θα επηρεαστεί υπερβολικά από, το, τα λόμπι και θα, ακούστη, θα εισακούεται η φωνή του πολιτή. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε πιο πολύ διαφάνεια στα θέματα διαπραγματεύσεων όπως οι πολύ αμφιλεγόμενες ε, διαπραγματεύσεις για το TTIP. Σήμερα βέβαια αυτό είναι λίγο εκτός θέματος με τις ε, ε, αμερικανικές εκλογές κατά πάσα πιθανότητα είναι πλέον τμήμα του παρελθόντος το TTIP, αλλά σίγουρα έχουμε λάβει πάρα πολλά αιτήματα για διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διαπραγματεύση το εμπόριο. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε την πλήρη δημοκρατική δηλαδή, διαδικασία έλεγχου για όλους ε, τους κανονισμούς και όλες τις ρυθμίσεις και επίσης Υπάρχει το θέμα της ανησυχίας που θα σήμαινε η έλλειψη Ευρώπη σε πολλά σημεία νομοθεσίας, γιατί πολλές αναφορές έχουν να κάνουν με ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη, όπου η έλλειψη νομοθετικής ή η λυπής εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας τελικά έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ανομοιογενές ε, μια ανομοιογενής εικόνα και ο πολίτης να έχει την αίσθηση ότι δεν υπερασπίζεται κανείς τα δικαιώματά του. Είναι σημαντικό λοιπόν να εισακουστεί η επιθυμία μας προκειμένου να καταλάβουμε ποιο είναι το κόστος πραγματικά του να μην υπάρχει Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί υπάρχει κόστος του να μην λαμβάνονται κάποιες συλλογικές δράσεις για τον πολίτη και αυτό το βλέπουμε τακτικά εμείς. Και πάντα καταλήγουν οι πλέον ασθενείς να πληρώνουν την ύφη. Θα υπάρχουν ε, λοιπόν και θα κατευθούν μια σειρά από τροπολογίες, ελπίζουμε να τις λάβει υπόψη ο εισηγητής και προσβλέπουμε στη συνεργασία με τον εισηγητή και να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση η οποία τελικά θα λεφτεί υπόψη από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και θα καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση τελικά. Σας ευχαριστώ λέει και Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ αλλά δεν είναι συνταγματικών υποθέσεων η καθήλυνα αρμόδια, είναι η γιούρη νομικών υποθέσεων. Η δική μας γνωμοδότηση παρόλα αυτά ελπίζω να ληφθεί υπόψη και από την γιούρη. Ο εισηγητής. Μεγάλη έμφαση στην ψήφιση της έκθεσης για τον Διάμεσο διαμεσολαβητή και μου διέλαθε ότι έχουμε και τη συζήτηση αυτής της σημαντικής ε, ε opinion. Ε, Καταρχά να πω ότι θα ακούσω βεβαίως και τους υπόλοιπους ε, ε, σάντο ε, και τις παρατηρήσεις τους, ώστε να πάμε σε μια ισορροπημένη έκθεση, η οποία θα απηχεί όλες τις απόψεις για να μπορέσει να έχει τη μεγαλύτερη στήριξη. Η καλύτερη νομοθέτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως έχει δύο πλευρές, έχει την τυπική και την ουσιαστική. Σε επίπεδο ουσιαστικής νομοθεσίας θα πρέπει να έχουμε μια νομοθεσία κοινωνικά ισορροπημένη. Αυτό άλλωστε επισημαίνεται και στην ε, γνωμοδότηση στην πρώτη παράγραφο, διότι έχουμε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια νομοθεσία η οποία πολλές φορές δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Ε, δεν βοηθάει στην απασχόληση και φυσικά οδηγεί και ε, πολλές φορές ε, ε, σε εντάσεις ε, και φυσικά σε λήψη αποφάσεων οι οποίες δεν ε, στηρίζουν τα συμφέροντα της πλειοψηφία των ίδιων των πολιτών. Άρα λοιπόν το πρώτο στοιχείο είναι η κοινωνικά ισορροπημένη νομοθεσία. Το δεύτερο έχει σχέση με την απασχόληση πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες ενισχύουν την απασχόληση και ενισχύουν τα κοινωνικά δικαιώματα, διότι βρισκόμαστε σε μια φάση εκτεταμένης ανεργίας και υποαπασχόλησης, σε μια φάση σημαντικής κοινωνικής φτώχειας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα λοιπόν η νομοθεσία πρέπει να ενεργεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να κλείνουν οι πνιγές της ανεργίας και των μεγάλων ανισοτήτων. Και αυτό επισημαίνεται στην παράγραφο 4. Το επόμενο θέμα έχει σχέση με την περίφημη TTIP, δηλαδή την γνωστή συμφωνία, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη δεν συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο στις πολυεθνικές, επίσης ε, καταργεί ουσιαστικά τα, ε, τα δημόσια αγαθά, δημιουργεί ένα δικαστικό ή παραδικαστικό σύστημα που αμφισβητεί την, ε, το ίδιο το δικαιοδοτικό σύστημα των κρατών μελών και διαλύει την αγροτική οικονομία. Βεβαίως ε, με τις τελευταίες εξελίξεις και την εκλογή Τραμπ είναι πιθανό να μην προχωρήσει αυτή η συμφωνία και αυτό είναι ευχάριστο πιστεύω για τους λαούς της Ευρώπης και ιδίω για τους Έλληνες πολίτες. Ε, αναφερόμαστε όμως στο ζήτημα της νομοθεσίας σε σχέση με την TTIP, δηλαδή την εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων, Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των ίδιων των ε, ε, ευρωβουλευτών και φυσικά της ίδιας της ε, ευρωπαϊκής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων όσων δηλαδή πλήττονται από αυτή την συμφωνία. Επίσης, ορισμένα άλλα θέματα έχουν σχέση με την συνεργασία του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, διότι είναι τα δύο νομοθετικά σώματα, πρέπει να έχουν μια καλή συνεργασία μεταξύ τους, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς ως Ευρωβουλευτές, ως το σημαντικό ε, σώμα, νομοθετικό σώμα της Ένωσης, να παίζουμε το ρόλο μας και να συμβάλλουμε στην ευημερία των ίδιων των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Ε, και το επόμενο θέμα και με αυτό κλείνω είναι ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων ο οποίος είναι σημαντικός αλλά θα πρέπει ε, να υπάρχει αν θέλετε μια ε, ρύθμιση τέτοιου τύπου ώστε οι εμπειρογνώμονες πραγματικά να συμβάλλουν ε, στην καλύτερη νομοθεσία και να φύγουμε από την αντίληψη περί αποπολιτικοποιημένης νομοθετικής διαδικασίας ότι όλα δήθεν είναι θεσμικά και ότι δεν ε, ασκούμε πολιτική. Ασκούμε πολιτική, παίρνουμε συγκεκριμένες αποφάσεις που σημαίνει συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές επιλογές. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία της ε, ε, έκθεση. Άκουσα με ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις από την Σάντο Ραπορτέρ ε, του S&D. Θα ακούσω και τις υπόλοιπες παρατηρήσεις από τους συναδέλφους. Ε, είμαι ανοιχτό να δούμε και τις τροπολογίες οι οποίες θα κατατεθούν και να καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία να είναι ισορροπημένη και αποδεκτή ε, κατά το δυνατόν από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. And now the floor goes to Peter Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν έχω να κάνω πολλές ε, παρατηρήσεις, τα έχουν πει ήδη σκιώδες εισηγητές. Πιστεύω πως η γνωμοδότηση είναι αρκετά λεπτομερής και θα έπρεπε να τη λάβει υπόψη η Ερμόδια Επιτροπή. Συνήθως διαπιστώνεται μία ανάγκη για αλλαγή, τροποποίηση της νομοθεσίας και ε, νομίζω πως ε, η Επιτροπή μας και το έργο της υποτιμάται γενικότερα. Εμείς ε, ακούμε τις φωνές των πολιτών για το τι δεν λειτουργεί. Γι' αυτό λοιπόν... Καταρχά, θα επιθυμούσα μια καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη μορφή ενό επικοδομητικού διαλόγου έτσι ώστε να καταφέρουμε μαζί να διαπιστώσουμε τι ε, συμβαίνει, τι δεν πάει καλά, εάν υπάρχει συμμόρφωση ή όχι προς την νομοθεσία, τι πρέπει να αλλάξει ε, και να διαπιστώσουμε εάν εν τέλει υπάρχουν λάθη που πρέπει να διορθωθούν στη νομοθεσία. Μετά, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, ε, να βελτιωθεί η διαφάνεια. Συνήθως παρατηρούμε τελευταία μία αυξανόμενη ε, μια αυξανόμενη επικριτική διάθεση των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω πως ε, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και να το διορθώσουμε. Από την άλλη, να φροντίσουμε να διατηρήσουμε τις ισορροπίες σχετικά με τη διαφάνεια και να μην ξεχνάμε πως δούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και πρέπει να ακούμε τη φωνή των πολιτών. Πέραν αυτών να πω πως χαίρομαι ότι ο εισηγητής κατάφερε να συντάξει μια περιεκτικότατη γνωμοδότηση και πιστεύω πως μαζί με καλή συνεργασία θα καταλήξουμε σε μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Τουλάχιστον το ΕΛΚΑ έχει ε, ένα πάρα πολύ ε, θετικό πνεύμα, πνεύμα συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ, Πίτερ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ομιλητή που ζήτησε το λόγο, γι' αυτό λοιπόν νομίζω πω μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη κυρία Μαριά. Α, θέλετε το λόγο ξανά. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω του συναδέλφους. Άκουσα τι παρατηρήσει για την ε, γνωμοδότηση αυτή. Θα τις λάβω υπόψη, περιμένω τις τροπολογίες και θα ήθελα να ζητήσω ξανά συγγνώμη από του συναδέλφους γιατί ε, Είχα δώσει μεγάλη έμφαση προηγουμένως στην έκθεση για τον Ombudsman προκειμένου να περάσει και έτσι μου είχε, ε, δεν είχα δώσει ε, ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της γνωμοδότησης που πρέπει να συζητήσουμε. Ε, να με συγχωρείτε πολύ για την αριθμία η οποία προκλήθηκε στη συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο σημείο 15. Το σημείο 15 να σας ενημερώσω πώς ακυρώνεται, διότι ακυρώθηκε η διερευνητική αποστολή, η οποία ακυρώθηκε διότι υπήρχαν μέλη της Επιτροπής που ζήτησαν να γίνει, παρόλα αυτά δεν ε, βρέθηκαν εκεί την ώρα που έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ήρθαν. Θα επανέλθω όμως στο θέμα αυτό κατά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Όμως, Έγινε μια διερευνητική αποστολή και είναι στο σημείο 16 η διερευνητική επίσκεψη στη Σλοβακία που ε, έλαβε χώρα στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή με πολλά και ενδιαφέροντα ευρήματα. Νομίζω πως έχετε όλοι λάβει το σχετικό έγγραφο. Ήταν Τη Δευτέρα η προθεσμία αποβολή τροπολογιών. Όσες υποβλήθηκαν συμπεριλήφθηκαν στο κείμενο και τώρα τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να υποβάλουν τροπολογίες στις συστάσεις. Να το τονίσω αυτό, στις συστάσεις και όχι στο κείμενο του σχεδίου έκθεσης. Και να υποβάλουν τις τροπολογίες τους στην αγγλική γλώσσα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, την επόμενη Τρίτη δηλαδή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να υποβάλουν τις τροπολογίες συμπληρώνοντας το έντυπο που τους διανεμήθηκε από τη Γραμματεία. Στις 28 και 29 Νοεμβρίου θα ε, ψηφίσουμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής και θα μεταφραστεί το κείμενο στα Σλοβάκικα και σε όποια άλλη γλώσσα ζητήσουν τα μέλη. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για την έκθεση, εφόσον όλοι την έχετε διαβάσει θεωρώ, να Επισημάνω όμως ότι η σύσταση που έχω για σας είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις ε, τροπολογίες της συστάσεις να είναι στις... Στις 15 Οκτωβρίου, λέει η Πρόεδρος, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για την ψηφοφορία. Νοεμβρίου, Νοεμβρίου με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. 15 Νοεμβρίου. Αυτά λοιπόν για αυτό το σημείο και ας προχωρήσουμε στο σημείο 17. Αναφορά 1049 κάθετος 2015 από τον την LL με αρκετές υπογραφές σχετικά με την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Πού δω πού. Ο αναφέρον, η αναφέρουσα είναι εδώ. Και η γραμματεία της Ιταλικής Επιτροπής με το όνομα New Deal for Europe είναι επίσης παρούσα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω αμέσως το λόγο στους αναφέροντες για πέντε λεπτά το πολύ. Παρακαλώ. Noi promotori <clears throat> Εμείς ε, οι αναφέροντες με βάση το New Deal for Europe είμαστε πεπισμένοι ότι για να υπάρξει εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρώπη θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα δεδομένα που απορρέουν από την εφαρμογή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας μετά από πολλά χρόνια λιτότητας δίνουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας όμως δυστυχώς η περικοδότηση είναι ανεπαρκής για να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τα προβλήματα της ανεργίας, γιατί μιλάμε για 20 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις νέες προκλήσεις της μετανάστευσης και της εξωτερικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται άλλες πηγές ε, πόρων, διότι το 1 τρίτο των κρατών μέσα στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας μπορούν ε, να προωθήσουν ζητήματα που αφορούν το θέμα του χρηματοπιστωτικού φόρου έτσι ώστε να, αντισταθμιστούν, ε, να αντισταθμιστεί η βλάβη που έχουν υποστεί οι πολίτες. Δεύτερον, ε, ένας ε, φόρος για το διοξίδιο του άνθρακα έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε και τα ορυκτά καύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη και το χαμηλό κόστος του πετρελαίου. Επίσης, μπορούμε να φτάσουμε σε ε, ευρωομόλογα έργου μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και έργων. Επίσης, στα πλαίσια της ποσοτικής ε, χαλάρωσης θα πρέπει να δράσουμε άμεσα, όπως επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ατζέντα. Έχουμε να κάνουμε με την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και την ε, εργασία του Μάριο Μόντι μέσα στα πλαίσια της, του Ανώτατου Συμβουλίου για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών διαδικασιών. Το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο μπορεί να τα καταφέρει και να βοηθήσει στο να αρθούν τα προσκόμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει μία άποψη για την αναφορά μας και θα ήθελα να πω ότι επειδή ορισμένα κράτη αντιτίθενται στην αύξηση των ιδίων πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού, μία ομάδα κρατών μελών μπορεί να ζητήσει την αύξηση των ιδίων πόρων μέσα στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας. Αυτό το στοιχείο δεν το λαμβάνει υπόψη η Κομισιόν. Το αγνοεί πλήρως. Αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ 10 κρατών μελών για έναν ε, φόρο ως προς τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μαζί και με το φόρο ε, τον, φόρο για τη χρήση άνθρακα και ορυκτών καυσίμων θα μπορέσουμε να προβάλλουμε στρατηγικές επενδύσεις με τις συνεργαζόμενες χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους εθνικούς πόρους που θα μπορέσουν να χορηγηθούν στον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό για την ανάκαμψη των χωρών μας. Θα ήθελα να τονίσω και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει έκδοση ευρωομολόγων έργου και αυτό εξαρτάται από αντίστοιχους, αυτό αντισταθμίζεται και από αντίστοιχους πόρους, δηλαδή μιλάμε για 30 δις και 50 δις αντιστοίχως από αυτούς τους δύο φόρους. Για να φτάσουμε και στην έκδοση ευρωομολόγων. Θα ήθελα να πω ότι η αναφορά δεν είναι προσωπική μου πρωτοβουλία. Μιλάμε για μια εκστρατεία New Deal for Europe που έχουν προωθήσει 10 επιτροπές σε 10 κρατη όπου συμμετέχουν και 68 ΜΚΟ καθώς ε, και 13 συνδικάτα, 126 δήμαρχοι μεταξύ των οποίων του Παρισίου της Λίλης, της Λιών, της Ρώμης και του Τωρίνο. 73 ε, ευρωβουλευτές επίσης είχαν συμμετάσχει και πέντε από τους 6 υποψηφίους για την Προεδρία του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και αντίστοιχα πολιτικά κόμματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προσώπου της να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Μάουρα από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού του τμήματο ε, που διαχειρίζεται ίδιου πόρου και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του αναφέροντε για την ε, παρουσίαση και να πω πω ήδη λάβατε την ε, απάντηση τη Επιτροπή τον Ιούνιο. Σε γενικέ γραμμέ να πω πω καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία σα που ήταν πολύ εμπνευσμένη. Στο μεταξύ, να πω πως οι προτάσεις για την ενδιάμεση αναθεώρηση έχουν ήδη υποβληθεί και μάλιστα συμπεριλαμβάνουν αρκετά από τα θέματα τα οποία θίξατε στην αναφορά σας. Για παράδειγμα, τη συνέχιση του ΕΦΣΥ ή τη συνέχιση της στήριξης στις πολιτικές προτεραιότητες που αφορούν τις θέσεις απασχόλησης, την ανάπτυξη και το μεταναστευτικό και προσφυγικό. Δεδομένων λοιπόν των περιορισμών ε, που υπάρχουν στα όρια του υφιστάμενου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους ε, μηχανισμούς του. Τώρα, σε σχέση με τους ε, ίδιους πόρους, να πω ότι καταρχάς γνωρίζετε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στην ομάδα υψηλού επίπεδου για το θέμα αυτό και να πω πως εξετάσαμε με μεγάλη προσοχή τις προτάσεις. Η ενισχυμένη συνεργασία δεν είναι κάτι που αγνοούμε. Αν θυμάστε καλά, μάλιστα, η πρόταση αυτή προέρχεται και από τους ε, ίδιους ε, πόρους. Όμως, ε, τα έσοδα από τους ίδιους ε, πόρους ε, δεν βρίσκονται εντός των ε, διαπραγματεύσεων. Ακόμα και από την ομάδα που τα διαχειρίζεται. Ωστόσο, ας μην αποκλείσουμε τίποτα, ας μην κρίνουμε εκ των προτέρων, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά να πω πως προς το παρόν νομικά τουλάχιστον δεν έχουμε κλείσει καμία πόρτα. Όλα είναι πιθανά. Γι' αυτό λοιπόν η απόφαση για τους ίδιους πόρους στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης ε, δεν είναι κάτι προς συζήτηση προς το παρόν. Θα το δούμε μακροπρόθεσμα, θα το εξετάσουμε στα πλαίσια του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Να σας πω πως ε, ήδη το 2017 θα μπούμε στη διαδικασία προετοιμασίας. και θα συζητηθούν οι προτεραιότητες των δαπανών, θα συζητηθεί η δομή του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, η δομή των εσόδων και όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν τη βάση του προγραμματισμού για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν να είστε σίγουροι ότι οι προτάσεις σας θα συμπεριληφθούν στις ε, προετοιμασίες μας. Και να πω και κάτι άλλο ότι σε ό,τι αφορά τις θεσμικές διαδικασίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ε, ενεργά όχι μόνο για τις δαπάνες αλλά και για τους ίδιους πόρους και τα έσοδα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ε, έχει αναφερθεί από πολλά εξέχοντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ε, συζητήσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό να είστε σίγουροι δεν σας αγνοούμε. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Πρώτη ομιλήτρια, κυρία Ρούσκα Καμπεσόν. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά γιατί νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να δούμε ποια είναι η άποψη και άλλων επιτροπών και των προϋπολογισμών καθώς και τις απασχόλησης που υποστηρίζουν αυτή την ιδέα. Δέχομαι τις θέσεις του αναφέροντα και χαίρομαι και την ανταπόκριση της Κομισιόν. Όπως είπε και ο αναφέρον, η οικονομική κατάσταση είναι δεινή, αντιμετωπίζουμε πολλές ε, κοινωνικές προκλήσεις, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις χώρες που γνωρίζουν μία δυσχερή κατάσταση. Πιστεύω ότι η ενισχυμένη συνεργασία θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία και όπως σας είπα θα πρέπει να ζητήσουμε και την υποστήριξη άλλων επιτροπών για να συνεργαστούμε. Αυτά. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές στον κατάλογο, κάτι το οποίο με εκπλήσει. Ο Πέτερ. Ναι, να πω πως... Ε, καταρχάς δεν ζήτησα το λόγο γιατί συμφωνώ απόλυτα με την ε, κυρία Ρούσκα Πεσόν. Εδώ τι συμβαίνει. Τα κράτη-μέλη, κατά ένα περίεργο τρόπο, ζητούν περισσότερη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουν ξεχάσει τις ίδιες τους τις υποχρεώσεις, έχω την αίσθηση. Ε, στη Γερμανία, ξέρετε, όταν ζητάς κάτι πρέπει και να το πληρώσεις ε, και να πω ότι ήδη οι πόροι σίγουρα είναι ένα πρόβλημα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αναφέροντες μας έδωσαν πάρα πολύ τροφή για σκέψη, πρέπει να πω. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα, πρέπει να εξετάσει το πού πρέπει να διατεθούν πόροι, αλλά να δει κιόλας και πώς θα λύσει το πρόβλημα των εσόδων. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αναφορά σας, να μας εμπνεύσει για τις ε, περαιτέρω συζητήσεις μας. Και να κρατήσουμε σίγουρα όλες τις πόρτες ανοιχτές. Ε, υπάρχουν βέβαια και πολλά θετικά. Να πω ας πούμε ότι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Πιστεύω πως... Ε, όταν βρισκόμαστε στο χείλο οικονομική καταστροφή μα έχουν κολλήσει στον τοίχο πω ένα, ένας φόρο ενδεχομένω να έλυνε τα προβλήματά μα. ή τουλάχιστον ένα μέρο αυτών. Γι' αυτό λοιπόν ε, είμαι απόλυτα και 100% υπέρ των αναφορών. Πρέπει να υπάρχουν αναφορέ έτσι ώστε εμεί να μπορούμε να εντοπίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην ομαλή λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπαθούμε να τα λύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμεί e eh, θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Θεωρούμε ότι υπάρχουν ε, πολλές δυνατότητες, γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αναφορά για να παραμείνει ανοιχτή η διαδικασία και να ζητήσουμε και την άποψη άλλων επιτροπών και προωθώντας και συνομιλία με την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη για αυτά τα θέματα που είναι αποφασιστικής σημασίας για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες, συμμερίζομαι τις ανησυχίες τους και θεωρώ ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια για να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και το 2017 να δούμε πώς θα έχει εξελιχθεί η συζήτηση. Ωραία. Εξαιρετικά ε, Γιώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ σε σχέση με τα ευρωμόλογα έργου νομίζω ότι μπορούν να ε, ε, εκδοθούν τη στιγμή που τηρούμε μία ισορροπία. Εάν μπορέσουμε ε, δηλαδή να προωθήσουμε το πολιετές και να αυξήσουμε τους ίδιους πόρους, τότε θα πρέπει να καταβληθεί η απόδοση κεφαλαίου σε αιτήσια βάση. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή αναμένοντας την αντίδραση της Επιτροπής έτσι ώστε να γίνει αύξηση των ιδίων πόρων για να μπορέσουμε να εκδώσουμε τα ευρωομόλογα και βεβαίως να υπάρξει και μία αύξηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κάλβες. Σα Σας ευχαριστώ. Ποιες γλώσσε γλώσσες να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω. Όποια θέλετε από τις 24 επίσημες. Ε, αλλά επειδή μίλησε ο συνάδελφο ε, σε καλά αγγλικά, Α, νόμιζα ότι μπορούσε να μιλήσει ισπανικά. Όχι, γιατί γλώσσα θέλετε. Τώρα που μίλησε αγγλικά, τον κατάλαβα τον συνάδελφο για πρώτη φορά. Εγώ απλώς θα ήθελα να πω εξ ονόματος των φιλελευθέρων, γιατί βλέπω ότι είμαι μόνος εκτός από την ε, πρόεδρο που πρέπει να τηρήσει ουδετερότητα. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει και το ρόλο του Κοινοβουλίου που νομοθετεί και έχει και ένα ευρωπαϊκό υπόβαθρο. Δεν αφορά μικροδιενέξεις τοπικού χαρακτήρα. Είναι μία πολύ στεναρή πρόταση στην οποία θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια. Θα πρέπει η ΠΕΤΗ να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανοίξει αυτή η συζήτηση ε, βεβαίως υποστηρίζοντας αυτή την κίνηση θα πρέπει να δούμε ποιες αποχρώσεις και θέσεις προβάλλει κάθε πολιτική τάση. Όμως είναι μια πρόταση για μια καλύτερη Ευρώπη, για μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη και πιστεύω ότι θα πρέπει πρέπει να συγχαρούμε τους αναφέροντες και η ΠΕΤΗ θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί και εμείς θα την υποστηρίξουμε. Ωραία. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο. Όχι. Θα ήθελα να σας πω ότι θα έχετε λάβει μία επιστολή από τον πρόεδρο Τσέκον Ζητήσαμε και τη συνεισφορά της Επιτροπής Απασχόλησης για αυτό το θέμα και η Επιτροπή Προϋπολογισμών ήδη μας απάντησε το Σεπτέμβριο. Συμφώνησαν ότι χρειάζεται κοινοβουλευτική συνεργασία σε αυτά τα θέματα και μιλούν για την διαθεσμική διάσκεψη του Σεπτεμβρίου για την μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμμετείχαν και τα εθνικά κοινοβούλια και συζήτησαν θέματα ε, δημόσιας κρατικής χρηματοδότησης και βεβαίως το θέμα των ιδίων πόρων. Επίσης αναφερθήκαμε στο ψήφισμα του Ιουλίου για την περίοδο 14-20 του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου καθώς και την αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων. Και πραγματικά ε, οι δύο φόροι που προβάλλουν οι αναφέροντες έχουν πραγματικά νόημα θα πρέπει να τους εξετάσουμε. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών επίσης τόνισε ότι η αναθεώρηση των ιδίων πόρων δεν πρέπει να συνδέεται με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να αλλάξει το, ο κανονισμός ιδίων πόρων. Τώρα, η επιστολή αυτή που είναι άκρος ενδιαφέρουσα, ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη την υπογράφει, πρόεδρος της ΕΚΟΝ, αναφέρει τα εξής. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ ακόμα δεν έχει εγκρίνει και λάβει τελική θέση επί της πρότασης αυτής, αλλά ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουμε μία φορολογική πολιτική και ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ε, δεν υπάρχουν νομικές ε, αρμοδιότητες, αλλά η δημοκρατική λογοδοσία θα πρέπει να ισχύει σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, αναφέρει, θα διαβιβάσω αυτή την αναφορά και τα παραρτήματα στην ε, ομάδα διαπραγμάτευσης της ΕΚΟΝ και έτσι θα γίνουν περαιτέρω διαβουλεύσεις και θα μας ε, ενημερώσει σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τώρα τα γνωρίζουν αυτά οι αναφέροντες και θα ήθελα ο κύριος Τέρικα Μπράς να λάβει το λόγο. Thank you, Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε κι εσείς, πριν από λίγο, η διερευνητική αποστολή στο Ταράντο ακυρώθηκε, αναβλήθηκε. Υποτίθεται ότι θα ήμουν κι εγώ μέλο τη αποστολή αυτή. Ναι, δεν το συζητάμε όμω αυτό τώρα, λέει ο πρόεδρο. Συζητάμε την αναφορά. Α, συγγνώμη. Νόμιζα ότι θα λένε να τελειώσετε και πριν τελειώσετε να αναφέρουμε και δύο λόγια, να πούμε δύο λόγια ε, για την ερευνητική επίσκεψη. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη και σα ζητώ συγγνώμη που σα διακόπτω. Α, ωραία, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα να δώσω το λόγο λοιπόν και πάλι στον αναφέροντα. Ή μήπω. Όχι, στον αναφέροντα. Να ακούσω τι έχετε να πείτε σε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και ενδεχομένω και σε αυτά που ανέφερε ο συνάδελφο από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν, γιατί όλοι εκτιμήσατε θετικά την πρότασή μας. Άρα το αίτημά μου είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να εξεταστούν διάφορες προτάσεις από τις αρμόδιες επιτροπές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογραμμίζω το γεγονός ότι υπάρχει ένα κίνημα από τη βάση που ζητά να υπάρχει υψηλότερη πρικοδότηση με ίδιους πόρους του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και Στα πλαίσια της Ευρωζώνης, των χωρών της Ευρωζώνης και μέσω ενισχυμένης συνεργασίας πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να γίνει ένα πρώτο βήμα το οποίο το 2020 θα οδηγήσει στην αύξηση των ιδίων πόρων του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μια απόπειρα να συνοψίσω. Καταρχάς, να στραφώ προς εσάς, ε, κύριε. Να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας και θερμότατα. Θα σας ευχαριστώ για την πολύ καλή συμβολή σας για την αναθεώρηση του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου. Και νομίζω ότι ως πολίτης της Ευρώπης μπορείτε να είστε περήφανος ότι επιτελέσατε το καθήκον σας με θαυμάσιο τρόπο με την αναφορά αυτή, γιατί καταφέρατε ήδη <coughs> να επηρεάσετε τις εργασίες που γίνονται για το θέμα αυτό. Έχει λεφθεί υπόψη ναι, η αναφορά σας, όχι μόνο από την Επιτροπή Αναφορών, αλλά και από την Επιτροπή Προπολογισμού από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Απασχόλησης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ίδια. Άρα, η αναφορά σας είναι στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Εργασίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό πραγματικά δεν είναι συνηθισμένο, ξέρετε. Μία αναφορά να καταφέρει να αλλάξει και να έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο σε τόσα πολλά επίπεδα. Σας ευχαριστούμε να σας ε, ε, διαβεβαιώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσα της ομάδας ε, υψηλού και ιδίων πόρων και μέσω του διαλόγου με τα Εθνικά Κοινοβούλια συμμετέχει συστηματικά στα ζητήματα αυτά τα οποία άπτεται η και θα συνεχίσουμε τις εργασίες βάσει τη συμβουλή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα βλέπω ότι φτάνουν σιγά σιγά και άλλοι συνάδελφοι πάνω που ήμουν έτοιμοι να κλείσω. Ναι, συγγνώμη, λέει, πρόεδρε, λέει ο κ. Λόμπος Αγγιλάρ. Ε, ε, συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά ιδιαίτερα εμείς που είμαστε, ε, δεν είμαστε μόνιμα μέλη της Επιτροπής ε, Αναφορών, έχουμε δυσκολίες να είμαστε στην ώρα μα γιατί πηγαίνουμε από τη μία συνεδρία στην άλλη. Αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, ναι, βεβαίω. Εγώ βλέπω τον αναφέροντα, ο οποίος γνέφει καταφατικά στο πώ συνόψισε τη συζήτηση. Να σα πω όμω ένα στοιχείο να σα αναφέρω. Σήμερα έχουμε χρόνο. Και όταν ο Χουάν Φερνάντο έρχεται στη συνεδρία είναι τιμή μου και χαρά να του δώσω το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. σα ευχαριστώ, Σεσίλια. Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να χαιρετήσω λοιπόν την παρουσία ανθρώπων οι οποίοι έχουν κινητοποιήσει όλες τους τις δυνάμεις και άλλους ανθρώπους έτσι ώστε να γίνει μια νέα συμφωνία για την Ευρώπη. Κάθε φορά που συζητούσαμε το θέμα αυτό, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και να καλωσορίσουμε τις ιδέες σας, τις ιδέες οι οποίες προτείνουν να συνδυάσουμε τα εφιστάμενα μέσα στα πλαίσια του σχεδίου Juncker έτσι ώστε να γίνει μια νέα συμφωνία για την Ευρώπη. Και να χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή θέλουμε μια δημοσιονομική πολιτική που να ευνοεί την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να σταθεί πάλι στα πόδια της οικονομία της Ευρώπης. Αλλά νομίζω πως για άλλη μία φορά βλέπουμε πάλι το ίδιο μοτίβο. Βλέπουμε κατάχρηση και δυστυχώς δεν βλέπω να έχουμε αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, αντί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για να έχει το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων νέους πόρους, για παράδειγμα μέσω του φόρου χρηματοπιστωτικών επενδύσεων, το φόρο για το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό που κάνουμε είναι να διαθέτουμε πόρους από αλλού, δηλαδή να κάνουμε ανακατανομή πόρων να παίρνουμε από το ένα ταμείο και να δίνουμε στο άλλο. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε και το κίνημα που ζητά μια νέα συμφωνία, ένα νέο New Deal για την Ευρώπη και νομίζω πως είναι αρκετά επίκαιρο, πιο επίκαιρο από ποτέ. Είναι μάλιστα τώρα μια ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να ζητήσει αύξηση του προϋπολογισμού για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, Να δημιουργηθεί ένα εργαλείο δηλαδή που θα δρομολογήσει αυτό το νέο New Deal για την Ευρώπη. Αυτό το είπε και ο ίδιο ο πρόεδρο ο Γιούνκερ. Είναι ουσιώδε, είναι αναγκαίο και συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια υπαρξιακή κρίση η οποία μας ζητά, απαιτεί μάλλον να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά θα ήθελα να ζητήσω η, η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή μέχρι να αναλάβει επιτέλους δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προτείνει μια εισαγωγή νέων πόρων ε, που θα διατεθούν για επενδύσεις ε, που θα δώσουν όθηση στην ανάπτυξη και να αυξήσει τους πόρους του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πάρω τώρα την ευκαιρία αυτή για να το τονίσω άλλη μια φορά. Είμαι ένας από τους υπέρμαχους της πρωτοβουλίας αυτής. Σε ευχαριστώ πολύ Σεσίλια που μου έδωσες το λόγο. Ε, ναι, λέει η πρόεδρος. Και εγώ θυμάμαι όμως τις εποχές που ήσουν εσύ πρόεδρος και ε, τα ίδια πράγματα που λέγω σε σένα. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Έλλη Σλάμ, η οποία θα μας μιλήσει για κάτι τελείως διαφορετικό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Σεσίλια δεν είναι τόσο διαφορετικό αυτό που θα ήθελα να πω. Έχει να κάνει με τη ε, δουλειά που κάνουμε για τη μεταρρύθμιση του φυστάμενου πλαισίου και θα ήθελα να συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα και να πω ότι σας ευχαριστώ για αυτή την αναφορά το New Deal για την Ευρώπη είναι ύψης της σημασίας, κάτι το οποίο υποστηρίξαμε κατά την προεκλογική μας εκστρατεία για τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι ε, αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις τους τελευταίους ε, τέσσερις μήνες ε, γνωρίσαμε την ψήφο υπέρ του Brexit και χτες το βράδυ, σήμερα το πρωί, γνωρίσαμε και τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος δρόμος για να καταστήσουμε κατανοητό στους πολίτες το τι σημασία έχει να υπάρχει μια ενωμένη Ευρώπη για αυτούς. Επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι ίδιοι πόροι. Μιλάμε για το φόρο άνθρακα και το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εμείς οι φεντεραλιστές Είμαστε πεπισμένοι ότι οι προκλήσεις αυτές είναι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες που δεν μπορούν να βρουν ε, λύση σε εθνικό επίπεδο. Τη στιγμή που ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει κοινέ λύσεις τις οποίες χρειαζόμαστε για το μεταναστευτικό και του αθέμητου ανταγωνισμού των ευρωπαϊκών κρατών και του του αυτού ανταγωνισμού χωρών που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την γεωπολιτική μας θέση στην παγκόσμια σκακέρα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει κοινέ απαντήσεις, αλλά παράλληλα θα πρέπει να γίνει με έναν προϋπολογισμό που είναι πολύ περιορισμένος. Δηλαδή στην Ιταλία λέμε ότι ένα αυτοκίνητο, μία Φεράρι, δεν μπορεί να λειτουργήσει με κινητήρα ενός Fiat Cinquecento. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι υπάρχει επίγον χαρακτήρας για την πραγμάτωση αυτού του σχεδίου πιστεύω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την ολοκλήρωση έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το χάσμα γενεών που υπήρχε στο παρελθόν. Μάλιστα. Ο κύριος Μπενιφέη. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Κυρία Βίξτρομ, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και εγώ να συνεχίσω στα Ιταλικά, μιας και έχουμε και τον αναφέροντα από την Ιταλία. Που ήταν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φιτρελαστικού Κόμματος, ε, Και ως Ευρωπαίος Ομοσπονδιστής ε, συμμετείχα σε αυτή την πρωτοβουλία για τους Ευρωπαίους πολίτες που ήταν ο πρόδρομος αυτής της αναφοράς την οποία υποστήριξα και σε μια προγενέστερη ακρόαση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή γιατί είναι ένα μέσο κινητοποίησης και συζήτησης για όλα τα θέματα που προανέφεραν συνάδελφοι, για τους ίδιους πόρους, για ένα βιώσιμο σχέδιο επενδύσεων και με νέους τρόπους χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι από πλευράς ε, Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, το θέμα αυτό θα πρέπει να προωθηθεί. Συμμετέχω και σε εκείνη την ε, Επιτροπή. Μας ενδιαφέρουν συστήματα οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μέσα στα πλαίσια και επιδομάτων ανεργίας στην Ευρωζώνη και το Ταμείο Εγγύηση για τους Νέους. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε και πέραν από το περιορισμένο σχέδιο Juncker. Το θέμα είναι επίκαιρο, η αναφορά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, γιατί τα θέματα που προωθεί δεν έχουν αντιμετωπιστεί διεξοδικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε και εμείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Θα πρέπει να κινηθούν οι κυβερνήσεις μας που δρούν περιορισμένα και με μεγάλη καθυστέρηση. Θα πρέπει να δοθεί μία όθηση και ένα κίνητρο που προωθώ ως Ευρωπαίος Φεντεραλιστής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λούτσο Λέβη και όλους όσους προώθησαν την αναφορά και την, επανέφεραν, την έφεραν εδώ ενώπιόν μας. Πρόκειται για μια κοινή πορεία και την οποία θα προωθήσουμε περαιτέρω χρησιμοποιώντας αυτό το σημαντικό μέσο για να παραμείνει ζωντανή η συζήτηση. Πρέπει αυτά τα θέματα να τα συζητάμε ανοιχτά και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για έναν επιπρόσθετο προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη, να αυξήσουμε τους ίδιους πόρους και να βρούμε έναν κοινό τόπο αντιμετώπισης όλων αυτών των ζητημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, είναι πολύ ωραίο να είσαι πρόεδρος, ξέρετε, όταν όλοι συμφωνούμε. Και αυτό συμβαίνει και αυτό το απόγευμα. Συμφωνούμε όλοι, όλοι συνεισφέρουν, είναι εκπληκτική η δουλειά μα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες, να σας πω πως μπορείτε να επιστρέψετε στην Ιταλία με την αίσθηση ότι έχετε συνεισφέρει ως πολίτης σημαντικά σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα θεσμικά ομάδα της Ευρώπης. Και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, που δεν συμβαίνει συχνά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και καλή επιστροφή στην πατρίδα σας. Συνάδελφοι, έχω όρεξη σήμερα. Πάμε για καφέ, διάλειμμα. Ε, τι λέτε. Ε, κύριε Τερικάμπρας, θέλετε να πείτε κάτι. Είστε τόσο γενναιόδοροι μαζί μου και το εκτιμώ αυτό βαθύτατα. Σας ευχαριστώ. Να ζητήσω συγγνώμη για την προηγούμενη παρέμβαση που έκανα, γιατί άρχισα να έρθω. έρθω. Ήμουν σε μια τελείω διαφορετική επιτροπή και δεν ήξερα τι ακριβώ γίνεται, γι' αυτό συγγνώμη. Να περάσω τώρα στο θέμα. Ανακοινώσατε ότι ακυρώθηκε η διευνητική αποστολή στο Ταράντο. αναβλήθηκε, ακυρώθηκε. Να πω ότι λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι που τελικά ακυρώθηκε. Ναι, σε εσά μιλώ. ναι, ναι, με συγχωρείτε. Να πω τα εξή, πολύ σύντομα. Ότι θεωρώ πως είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτή την επίσκεψη, που δεν κατάφεραν να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι. και να πω ότι μας ανακοινώθηκε η ακύρωση της επίσκεψης λίγο πριν. Και εμείς που ήμασταν εκεί και ανυπομονούσαμε να πάμε, βρεθήκαμε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Με μεγάλη μας έκπληξη. Πιστεύω πως αυτό δεν είναι καλό για τη φήμη της δικής μας Επιτροπής και ιδιαίτερα για εκείνους που περίμεναν αυτή τη μέρα. Πώς και πώς. Ε, να, θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποια άλλη ημερομηνία για να γίνει αυτή η επίσκεψη που ακυρώθηκε. Σας ευχαριστώ. Ε, και εγώ λυπάμαι για την ακύρωση. Σημερίζομαι την αγανάκτησή σας. Αλλά είναι πολύ άσχημη εικόνα, ξέρετε, που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν πηγαίνει κάπου με ένα μέλος, δύο ε, μέλη και είμαστε τόσο λίγοι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προγραμματίσει να πάμε στο Τάραντο τη Ιταλία ε, από τις 2 στις 4 Νοεμβρίου. Θα ήσασταν στην αποστολή εσείς κύριε Τερικάμπρας και η κυρία Πιτέρα και επίσης κάποια άλλα μέλη, ο κύριος Κονσολίνο αν δεν κάνω λάθος και η κυρία Εύα το και ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να πάμε στο χαλιβουργείο της Σίλβα και στις εγκαταστάσεις του Ταράντο. Και είναι πραγματικά κρίμα το ότι μας ακύρωσαν τελευταία στιγμή πολλά μέλη. Εάν ακυρωθεί κάποια επίσκεψη σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων εβδομάδων, να ξέρετε πρέπει να πληρωθούν πολύ να πληρωθούν οι διερμηνείς. Και αν οι φορολογούμενοι μάθαιναν το κόστος αυτών των ακυρώσεων, τι θα γινόταν. Θα τα πούμε αυτά στους συντονιστές αργότερα, αλλά θέλω να τονίσω πως χρειάζεται πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας. Δεν μπορούμε να σπαταλάμε τα χρήματα των φορολογούμενων και να δίνουμε την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι δεν ενδιαφέρεται. Είναι εξίσου άσχημη η εικόνα που δίνουμε με μία κύρωση, είναι εξίσου όμω άσχημη και η εικόνα που δίνουμε όταν έρχεται ένα, ε, δύο ευρωβουλευτέ και μια ομάδα διερμηνέων. Συμφωνώ, λέει ο κ. Τερικάμπρα. Πλήττει την αξιοπιστία μα, ξέρετε, λέει ο πρόεδρο. Η, ε, η επιτροπή αυτή διέπεται από κανόνε και του κανόνε αυτού πρέπει να του ακολουθούμε όλοι. Αυτοί είναι κανόνες οι οποίοι προϋπήρχαν και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και με τους κανόνες των επιτροπών αποφάσισα ότι δεν είναι καλό να γίνει επίσκεψη με τα μέρη που ήταν παρόντα και δεν επιτρέπεται άλλωστε. Ναι, νομίζω πως έπρεπε να κυρωθεί αναγκαστικά γιατί δεν είχε νόημα. Το πρόβλημα ήταν ότι εξαφανίστηκαν τα μέλη της αποστολής αργά και σταθερά, αλλά δεν είχε μείνει κανεί. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε τα πράγματα πιο πολύ στα σοβαρά όταν διοργανώνουμε ε, τέτοιε αποστολέ. Και εγώ σα έστειλα αμέσω ένα μήνυμα. Σα είπα ότι συμφωνούσαμε να ακυρωθεί η αποστολή, γιατί δεν είχε νόημα να πάμε έτσι όπω ήμασταν. Αλλά σα ρωτώ, υπάρχει άλλη ημερομηνία που θα γίνει αυτή η αποστολή, διότι ξέρετε, μα περιμένουν εκεί μας περιμένουν πώς και πώς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ζητήσουμε από τους συντονιστές να θέσουν το θέμα στην ημερήσια διάταξη για να συζητηθεί εκ νέου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εγώ δεν μπορώ να αποφασίζω αυθαίρετα παρακάμπτοντας τους συντονιστές, ούτε η γραμματεία μπορεί να το κάνει αυτό. Πρέπει να ζητήσουν οι συνάδελφοι να συζητηθεί το θέμα στη συνεδρίαση των συντονιστών δεν προβλέπεται να συζητηθεί σήμερα στην ημερήσια διάταξη, αλλά θα συζητηθεί αργότερα από τη στιγμή που μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε να συζητηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανόνες. Ωραία, αυτό ρώτησα. Ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν και θα κάνουμε. Ναι, Μάρκερετ. Και εγώ θέλω το λόγο τώρα στη συνεδρίαση της Επιτροπής για να πω ότι αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι οι διερευνητικές αποστολές δεν μπορούν να συγκριθούν με τις αποστολές άλλων επιτροπών. Είναι ένα ε, αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας. Να σας πω και ότι εγώ η ίδια έχω συμμετάσχει σε αποστολές που ήμασταν μόνο δύο ευρωβουλευτές. Έχουμε πάει και οι πολίτες είδαν την αποστολή, είχαμε μια παρουσία, είδαν ότι κάποιος τους ακούει, δεν τους αγνοούμε. Και θέλω να το πω εδώ γιατί κάποτε είχαμε και μια γραμματεία η οποία είχε και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και μας στήριζε. Μας έλεγε ότι εντάξει, άμα δεν μπορεί να έρθει ας πούμε ο εκπρόσωπος του ΕΛ, καλά μην ακυρώσουμε να ζητήσουμε από κάποιον άλλο, από τους σοσιαλιστές, από κάποια άλλη πολιτική ομάδα να έρθει. Είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, αν δεν θέλει κάποιος να γίνει υποστολή, να μην ε, την κάνει, να φροντίσει να μην γίνει. Ε, ευχαριστώ. Ναι, και να πω εδώ πως ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τερικάμπρας γιατί είχε μείνει μόνος του. Αλλά ήταν εκεί. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να στείλουμε απόστολη ενός μόνο ευρωβουλευτή. Ε, άλλους συναδέλφους που πάνε αυτοπαγγέλτος. αλλά σας έδωσα το λόγο για να τα πείτε αυτά, γιατί ήσασταν ο τελευταίος που έμεινε. Αλλά να σας πω, θα το συζητήσουμε αργότερα. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών στις 5 ακριβώς, ούτε λεπτό αργότερα. Έχουμε πολλά να πούμε.